Okay. <laughs> Äh, äh, Κυρίες και κύριοι, αρχίζουμε την απογευματινή συνεδρίαση. Σας καλωσορίζω θερμά. Το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η έκθεση του κυρίου Παντσέρη για τα δασικά μηχανήματα. Είναι πολύ σημαντικό θέμα, όπως γνωρίζετε. Παρ' αυτά βλέπω ότι δεν είναι εδώ οι σκιώδες εισηγητής από τις ε, πολιτικές ομάδες. Θα σας πληροφορήσουμε όμως όταν έρθουν. Πρώτα δίνω το λόγο στον κύριο Παντσέρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως τα γνωρίζετε, ο στόχος της πρότασης είναι να προβλέψει μια σειρά από εναρμονισμένα πρότυπα για τα γεωργικά και δασικά οχήματα, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς χωρίς να χάσουμε το στόχο υψηλού επίπεδου περιβαλλοντικής προστασίας και, προστασίας και οδικής ασφάλειας για το εργασιακό περιβάλλον. Δεν θα σταθώ σε αυτό ιδιαίτερο, διότι τα συζητήσαμε και κατά τη διάρκεια της δημόσιας ακρόασης που διεξήχθη στις 12 Απριλίου σε επίπεδο τη επιτροπή μα και με την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε στις 30 Αυγούστου. Να ευχαριστήσω ευθύς εξ αρχή τους και εισηγητέ εισηγητές για τη συνεισφορά τους, τις διάφορες συναντήσεις που είχαμε και για την συνεργασία μας του τελευταίους μήνες. Συνολικά είχαμε 133 τροπολογίες, περισσότερες από τις οποίες δεν δημιουργούν δυσκολίες και τις οποίες θα τις σχολιάσουμε αναλυτικά στην επόμενη συνάντηση της συνεδρίας με τους κέντρους εισηγητές την επόμενη εβδομάδα. Ως προς την πρόσβαση στις πληροφορίες για τους ε, κατασκευαστές των ανταλλακτικών. Εδώ, πολλοί, πολλές τροπολογίες αναφέρονται στην απεριόριστη πρόσβαση στις πληροφορίες και την ανάγκη να προβλεφθεί ανάγκη η αναλογικότητα σε σχέση με τους εμπορευόμενους όγκους και τις συναλλαγές των εμπορευομένων. Εδώ μιλάμε και για τα οχήματα ή για τους μισθωτές. Επίσης χρειάζεται προστασία των σημάτων σε περίπτωση που αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι σημαντικό οι τεχνικές πληροφορίες να, να καλύπτουν τα τεχνικά σήματα, κάτι που ούτως ή άλλως το ισχύον, το κείμενο για τα κινούμενα με τα, μηχανοκίνητα μάλλον οχήματα καλύπτει και το εκτιμώντας 19 της οδηγίας 47 του 2007 το προβλέπουν, καθώς και για τα σήματα με προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας. Όσο για την απεριόριστη πρόσβαση, για να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση ως προς την πρόσβαση, για τους ανεξάρτητους εμπορευμένου, πρέπει ταυτόχρονα να καλύψουμε και τις ανάγκες των καταναλωτών, τα ζητήματα του θεμετού ανταγωνισμού και την περιβαλλοντική προστασία. Τέλος, και για τα οχήματα και όχι μόνο για τους μισθωτέ, θα μπορούσαμε να τα αποκλείσουμε από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, ιδίω τα οχήματα τη κατηγορία ΕΡΕ, των ρημουλκών και τη κατηγορία ΕΣΕ, που Αυτά ούτω ή άλλω δεν χρειάζεται να αποκλειστούν να συμπεριλαμβάνονται σε μια συνολική εξαίρεση. Για την πρόσβαση στις πληροφορίες θα μπορούσε να υπάρχει εδώ διακριτική μεταχείριση, όμως έχουν και ιδιαίτερο χαρακτήρα ε, η παραγωγή των ρημουλκών και των ρημουλκούμενων ε, μηχανικών εξαρτημάτων. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να βλεφτούν ειδικέ διατάξει με μικρότερες δεσμεύσεις, χαμηλότερες δεσμεύσεις για την παροχή πληροφοριών. Σε περίπτωση δηλαδή που παράγονται λιγότερε από 250 μονάδες θα μπορούσαν να παρέχονται πληροφορίες μόνο σε εκδοχή επιχάρτου. Εδώ δεν έχουμε έτσι κι ε, νομική υποχρέωση και δεν θα πρέπει να δυσχεραίνεται η υλοποίηση. Υπάρχει άλλωστε η Γενική Αρχή της Αναλογικότητας. Θα πρέπει λοιπόν να μελετήσουμε κατά πόσο είναι δυνατόν να πετύχουμε συμβαστική λύση σχετικά. Δεύτερο μεγάλο θέμα, το πεδίο εφαρμογή για τι κατηγορίε των οχημάτων. Πρώτη κατηγορία. Εδώ υπάρχουν διάφορε τροπολογίε που περιορίζουν το κείμενο σε σχέση με την κατηγορία U, δηλαδή τα μηχανήματα και τα κινητά μηχανήματα. Εδώ η αναφορά αυτή εξαλείφθηκε από το κείμενο γιατί θα χρειαστεί ad hoc διευθέτηση της κατηγορίας αυτής. Κάτι που ήδη έχει προβλεπτεί στην έκθεσή μας. Για τα μηχανήματα τα οποία δεν μπορούν να περιστραφούν γύρω από κάθε το άξονα. Εδώ υπάρχουν πολλέ τοπολογίε που ζητούν να μην ισχύει ο κανονισμό για τα μηχανήματα αυτά. Όμως τα ρημουλκούμενα μηχανικά εξαρτήματα ήδη είναι αντικείμενο έγκριση, ε, ανάλογα με τις συμβάσει μεταξύ των προμηθευτών. Οπότε δεν θεωρείται σκόπιμο να παραμείνουν αυτά τα μηχανήματα σε ένα κείμενο που δεν θα είναι σκόπιμο για τη συγκεκριμένη περίπτωση του Τώρα για, τα κατηγορία, για την κατηγορία C, σημεία 1 και 2, η ισχύουσα νομοθεσία ζητά ούτω ή άλλω, ανάλογα με τον τύπο οχήματο, να υπάρχει η έγκριση των ε, μηχανημάτων αυτών. Τώρα για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας στα πλαίσια της γενικότερης ρύθμισης και επειδή θέλουμε να πλουστεύσουμε το υπάρχον ε, ρυθμιστικό πλαίσιο για τους μισθωτές και επειδή θέλουμε να καλύψουμε καλύτερα τους υπάρχοντες κινδύνους ενώ ταυτόχρονα να υπάρχει δυνατότητα να καλυφθούν και αναδυόμενοι κίνδυνοι, όλα αυτά θα πρέπει να τα συνδυάσουμε και με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Γι' αυτό έχει προβληθεί μια σειρά αποτροπολογίες που αφορούν τη λειτουργική ασφάλεια, που καλύπτει και την προστασία στο χώρο εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα κείμενα. Δηλαδή τα μηχανήματα που, θα, που κάλυπταν οι οδηγίες που θα καταργηθούν μέσω του κανονισμού εφόσον εγκριθεί. Οι συστάσει αυτέ λοιπόν θα πρέπει να καλύπτονται στο κείμενο και θα πρέπει εδώ να είμαστε πολύ σαφεί. Ο κατάλογο του άρθρου 8 θεωρείται ένα κατάλογο διεξοδικό. Άρα, σε σχέση με τη λειτουργική ασφάλεια και εφόσον κάτι δεν θα περιλαμβάνεται στο άρθρο 8, δεν θα μπορεί κάτι να προσθεθεί εκτός άρθρου 8 με κάποιο παράρτημα ή με κάποιο άλλο τρόπο. Τώρα για, τη θέση για την ημερομηνία θέση σε ισχύ, για την ομολογοποίηση των ε, δασικών και γεωργικών οχημάτων. Εδώ είναι κρίσιμη η επιλογή της ημερομηνία, διότι μέχρι το 2014 θα έχουμε μια περίοδο νομοθετικής ε, δραστηριότητας, εντατικής δραστηριότητας, οπότε οι φορείς που θα ασχολούνται με την ομολογοποίηση θα πρέπει να καλύψουν ταυτόχρονα και τις απαιτήσεις της οδηγίας για τις εκπομπές. Άρα και η οδηγία για τα φρένα που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα και επειδή ενδεχομένω θα υπάρξει επικάλυψη όλων αυτών των νομοθετικών προτάσεων, θα πρέπει να βρούμε εμεί μια συμβαστική λύση που να διασφαλίσει ισορροπία μεταξύ τη απέτηση να δημιουργηθούν εναρμονισμένοι κανόνε και τι απαιτήσει των ενδιαφερόμενων φορέων, ώστε και την ομολογοποίηση να έχουν, αλλά και να μπορέσουν να ανασάνουν σε αυτή την εντατική περίοδο δραστηριότητα. Ένα τελευταίο σημαντικό πεδίο είναι πιο αντιφατική τυχή. τα επαγγελματικά οχήματα παντός εδάφου και οχήματα αναψυχή εκτός δρόμου. Εδώ δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ κρατών μελών και στο επίπεδο του Συμβούλου και δεν ξέρουμε αν αυτά τα οχήματα θα συμπεριφθούν στην κατηγορία L ή e T. Μιλάμε για τα οχήματα ATV και SBS. Εδώ μπορεί να μην μπορούν να ομολογοποιηθούν οχήματα με παρόμοια χαρακτηριστικά, με δύο ταυτόχρονε διαδικασίε ομολογοποίηση. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει λοιπόν προβλήματα ασφάλεια. Και μπορεί να μην υπάρχει ο κατάλληλο έλεγχο. Έπειτα, προ όφελο των Ευρωπαίων πολιτών και για καλύτερε περιβαλλοντικέ επιδόσει και λειτουργική ασφάλεια, είναι, θα πρέπει όλα αυτά να είναι σαφή. Εξάλλου, ω σήμερα δεν υπήρχαν σαφή τεχνικά κριτήρια για την κατηγοριοποίηση των οχημάτων αυτών που είναι αντικειμενικά και να επιτρέπουν να διακριθούν τα ATV από τα υπόλοιπα οχήματα. Η κατάσταση αυτή θα γίνει ούτω ή άλλω πιο περίπλοκη σε περίπτωση που τα οχήματα που φαίνονται να είναι παρόμοια τελικά ε, ε, υποπέπτουν, υποπέσουν σε δύο ταυτόχρονες διαδικασίες ομολογοποίησης. Αυτό πρέπει να το βρούμε με, με τους σκεώδεις εισηγητές και για παρόμοια οχήματα τα οποία δεν έχουν ε, εγκριθεί με μια κλασική διαδικασία μπορούν να περάσουν στην κατηγορία των μηχανημάτων. Θα θέλουμε λοιπόν να μην έχουμε μια ρυθμιστική, καταστροφική επέμβαση από την άποψη των, της ασφάλειας και του τύπου των οχημάτων. Επαναλαμβάνω ότι η κατηγοριοποίηση βάσει της χρήσης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Αυτή τη στιγμή ο ιδιοκτήτη μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το όχημα με τρόπο τελείω διαφορετικό από αυτόν που έχει προβλέψει ο παραγωγό. Αυτό συμβαίνει σήμερα και δημιουργεί μεγάλα προβλήματα ασφαλεία. Οι περιβαλλοντικέ ε, απαιτήσει ασφάλεια που προβλέπονται με τι διαδικασίε ομολογοποίηση τι δεν είναι επαρκή, ούτε μπορούν να καλύψουν ένα όχημα τόσο ταχύ όσο τα ATV. Άρα έχει αναφερθεί το γεγονό ότι η λύση να συμπεριλαμβάνουν να συμπεριλάβουμε όλα τα οχήματα ATV στην κατηγορία L ε, δημιουργεί προβλήματα και δεν είναι κατάλληλη. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε μια διαδικασία τέτοια, ένα ε, θεσμικό όργανο όπω το Ευρωκοινοβούλιο, που να είναι προ όφελο ολόκληρη τη κοινωνία. Όχι να βασιστούμε στι πιέσει μια συγκεκριμένη ομάδα ε, του πληθυσμού, δηλαδή των παραγωγών. Θα πρέπει εδώ να θεωρήσουμε να, να λάβουμε υπόψη μάλλον ότι κάποιε από τι αποφάσει μα μπορεί να ε, είναι αρνητικέ για κάποιον παραγωγό και θετικέ για κάποιον άλλο ή για την υπόλοιπη κοινωνία. Θα πρέπει επίση να δούμε ποιο είναι το κόστο τη ασφάλιση. Ε, το οχήματα ΕΛΕ πολλέ φορέ ε, πληρώνουν μεγαλύτερα τέλη από την κατηγορία T. Όμω αυτό δεν ισχύει για τα οχήματα επαγγελματική χρήση. Και τα ίδια τεχνολογικά μέσα μπορεί να αξιοποιούνται και στα ATV. Τα τεχνικά κριτήρια κατηγοριοποίηση, όπω ορίζονται στι τροπολογίε, μπορούν πολύ εύκολα να τροποποιηθούν εφόσον διαπιστωθούν παραβιάσει. Α θυμηθούμε τι τεχνικέ παρεμβολέ μπορούν να κάνουν οι ίδιοι ιδιοκτήτε των οχημάτων. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τέτοια τεχνικά κριτήρια τα οποία να μην μπορεί κανεί να τα πειράξει και να είναι και πολύ δαπανηρή οποιαδήποτε αλλαγή θέλει να κάνει κανεί στο όχημα. Θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφεί στι τεχνικέ ε, λεπτομέρειε και να μην επηρεάζεται η δυνατότητα ρημούλκησης ενός οχήματος, λόγου χάρη. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο αρμόζει τα ε, οχήματα ATV να συμπεριληφθούν στην κατηγορία αυτή, την L. Προφανώ δεν υπάρχει συνένεση για το θέμα αυτό, ούτε μια άποψη όλων, αλλά η συζήτηση αυτή θα πρέπει να γίνει στο επίπεδο τη διαδικασία πρόβλεψη νέων νομοθετικών κανόνων. Εν ολίγης, αυτά είναι τα βασικά σημεία που θα επεξεργαστούμε τις επόμενες Κυρίω κυρίως τη συνάντηση που θα έχουμε με τους σκεώδει εισηγητέ την ερχόμενη εβδομάδα. Είμαι πεπισμένος ότι πέραν των απόψεων που δικαιολογημένα μπορεί να είναι και διαφορετικέ, θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμβαστική λύση ώστε η Επιτροπή μα να καταλήξει σε ένα κείμενο που όλου λίγο πολύ να ικανοποιεί και να οδηγηθούμε σε ένα βασικό κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση για έναν τόσο σημαντικό τομέα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σίγητα και ευχαριστώ για την εκτενέστατη παρουσίασή σας. Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση είναι αρκετά τεχνική, ωστόσο έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στους κοιόδες εισηγητές ή τους αντιπροσώπους τους. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω μια ομάδα νέων ε, ομοσπονδιστών από την Κωνσταντζα οι οποίοι έχουν έρθει εδώ έχουν να δουν, για ε, να δουν πώς λειτουργεί η Ευρώπη, ποιος το κάνει, πώς το κάνει. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλωσορίσω και εύχομαι η σημερινή συνεδρία να μην είναι πολύ τεχνική για σας. Επίσης, θα ήθελα να χαιρετήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία βρίσκεται εδώ, την κυρία Χαχ, τον κύριο Αντρέα Βοσινής. Θα λάβατε και εσείς το λόγο στη συνέχεια. Επίσης τον κύριο Σφάμπ από το ΕΛΚ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι που βρίσκονται εδώ οι νέοι άνθρωποι από τη δική μου εκλογική περιφέρεια και ελπίζω να τους ε, φέρω κοντά με το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα με, τα, με τους ελκυστήρες ευχόμαστε η Κομισιόν να συνεργαστεί και να υπάρξει ένα καλό αποτέλεσμα. Η σκιώδη συγγήτρια ζητά συγγνώμη που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί και θα ήθελα να λάβω την ευκαιρία να σας ε, παρουσιάσω τις ε, θέσεις του ΕΛΚ για την για το θέμα αυτό. Αγαπητέ συνάδελφε Παντσέρη, πιστεύουμε, πιστεύουμε ότι η ρύθμιση των ε, γεωργικών μηχανημάτων θα μπορούσε να δεχτεί αρκετές βελτιώσεις. Έχουμε υιοθετήσει κάποιες τροπολογίες στο κεφάλαιο 16 όσον αφορά την πρόσβαση στην πληροφορία για τις ε, επισκευές. Ε, δεν ξέρουμε αν θα έπρεπε να παραμείνει αυτό στην ε, τροπολογία. Η κυρία Σαρτόρης, και η εισηγήτρια, έχει συντάξει αρκετές προτάσεις για τροπολογία και πιστεύω ότι η ομάδα μας θα επιθυμεί να εξετάσει αυτές τις τροπολογίες για να δούμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Πιστεύω όμως ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν έχει γίνει μελέτη αντικτύπου γι' αυτό και δεν υπάρχει λοιπόν επαρκή βάση, για να, ε, βάση της οποίας θα κάνουμε την πρότασή μας. Έπειτα, κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη γιατί έχω λίγο το λαιμό μου σήμερα, έπρεπε να αντιπροσωπεύσω πολλούς συναδέλφους. Έπειτα λοιπόν, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι η αρχή της ε, θέσης σε ισχύ της τροπολογίας είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ, αλλά το πότε είναι το σημαντικό για μας η έγκριση, οι νέες εγκρίσεις και οι υπάρχουσες εγκρίσεις είναι σημαντικό να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα. Ε, γι' αυτό και έχουμε συντάξει τις αντίστοιχες τροπολογίες. Αλλά πρέπει να τις συζητήσουμε και εδώ. Πιστεύω ότι η λύση για τα οχήματα κατηγορία L την οποία βρήκαμε είναι καλή βάση και ο εισηγητής έχει δουλέψει αρκετά στενά με τους εμπειρογνώμονες έτσι ώστε να το έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Κύριε Μπουζόη, ε, μου επιτρέπετε να δώσω πρώτα το λόγο στον συνάδελφό σας, ο οποίος πρέπει να φύγει. Τότε Έχω την τιμή να δώσω το λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής. Uh, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ uh, που ως πρόεδρος θα μπορέσετε να μας ελέγξετε όλους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Uh, λυπούμε διότι θα πρέπει να απουσιάσω σήμερα το απόγευμα, αλλά έχω ε, μια σημαντική ε, συνάντηση της Ευρωπαϊκής Κεραμοποιίας, αλλά πρέπει να βρίσκομαι εδώ τώρα, διότι είμαι σκιώδης εισηγητής και έχω καταθέσει τροπολογίες και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω, πρώτου χρειαστεί να φύγω. Συμφωνώ με τον Άντριο Σφάρ νομίζω ότι η βάση των όσων έκανε ο κύριος Παντσέρη είναι εξαιρετικά καλή και είχαμε την ευκαιρία ήδη να τον ευχαριστήσουμε διότι πρόκειται για μια πλήρη ε, και ενδελεχή ανάλυση και έχουμε εδώ πάρα πολλές βελτιώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία ε, λεπτομεριών πάνω στα οποία εργάστηκα. Θα ήθελα να αναφέρω κυρίως ένα σημείο ε, το οποίο σχετίζεται με την εργασία μας σχετικά με ε, τις ε, μοτοσυκλέτες. Νομίζω ότι τα οχήματα παντός εδάφους έχουν κάποιες διαφορές ε, ως προς τις απαιτήσεις, τις τεχνικές, τις ρυθμιστικές. Αλλά Νομίζω ότι αυτά τα δίκυκλα που χρησιμοποιούνται ε, και που πρέπει βεβαίως ε, να ακολουθούν τις ε, απαιτήσει ασφαλείας έχουν διαφορά με τις αγροτικά οχήματα ε, συζητήσαμε αυτές τις διαφορές και νομίζω ότι πάρα πολλοί ε, συνάδελφοι σκέφτονται ότι εφόσον έχουμε την ευχάριστη ευκαιρία να εξετάσουμε την οδηγία αυτή, ελκυστήρων ε, και μηχανημάτων ε, γεωργικών ταυτόχρονα και οχημάτων, ε, μια καλή κομψή λύση θα είναι να έχουμε μια ιδιαίτερη κατηγορία για τα ελαφρά αυτά οχήματα στην οδηγία για τα οχήματα αυτά που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς και νομίζω ότι μπορέσαμε να έχουμε έναν ορισμό που είναι αρκετά σαφής και ε, προσδιορίζει ε, τις απαιτήσει που για τα οχήματα, τα οδικά ε, που εμπίπτουν σε άλλη οδηγία. Βλέπετε ότι κατέθεσα ένα πακέτο τροπολογιών που συνυπογράφηκαν και από άλλους συναδέλφους και ελπίζω ο κύριος Παντζέρη να συμφωνήσει για αυτή την προσθήκη. Νομίζω ότι η χρήση ε, αυτών των οχημάτων, οι επαγγελματικοί οι χρήστες ε, θα ήσαν ικανοποιημένοι να έχουν την ίδια κατηγορία όπως η παραγωγή. Ε, και ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο κατά κάποιο τρόπο να γνωμοδοτήσει για να έχουμε μια ισορροπία ανάμεσα στις δύο κατηγορίες. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε και αν αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό θέμα για το οποίο ήθελα να συμπεριληφθεί. Υπάρχει και άλλες, υπάρχουν και άλλες τροπολογίες για ειδικέ κατηγορίες ελκυστήρων κυρίως για τους ελκυστήρες υψηλής ταχύτητας και θέματα σχετικά με τα συστήματα σταθερότητας για αυτούς τους ελκυστήρες και για την τροχοπέδη. Και έχουμε αυτές τις ελκυστήρες που είναι ικανοί για μεγάλη ταχύτητα. Θα θέλαμε να ενσωματωθούν στην βασική κατηγορία των οχημάτων. Γι' αυτό έχουμε ε, καταθέσει ε, κατά συνέπεια ορισμένε τροπολογίες για τον κύριο ε, Παντσέρη σχετικά με τα όσα είπε ο κύριος Σβάμπ για την πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες. Το εξετάζουμε αυτό εντελεχώς και επισύρω την προσοχή των συναδέλφων ότι παραγγείλαμε μία μελέτη και αυτό το βλέπετε στο φάκελο για την εξέταση ορισμένων θεμάτων. Νομίζω ότι η μελέτη ήταν ε, για μια βάση αλλά δεν οδήγησε σε ορισμένες ανησυχίες για τις προτάσεις. Μάλλον ε, θεώρησε ότι αυτό είναι ο καταλληλότερος τρόπος να προχωρήσουμε. Θα μελετήσω με ενδιαφέρον τις τροπολογίες του κυρίου Σβάμπ, αλλά νομίζω ότι για την ώρα θα πρέπει να ακολουθήσουμε την συμπρόταση που έχει η Κομισιό με ορισμένε διασφαλίσεις σχετικά με πληροφορίες για πάρα πολύ περίπλοκα μηχανήματα σε σχέση με μηχανήματα που μπορούν να επισκεφθούν επισκευαστούν με απλό τρόπο από επισκευαστές επιτόπιους. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα αυτό, αλλά για την ώρα δεν είμαι πεπισμένος ότι πρέπει ε, να υπερβούμε τα όρια ε, της εργασίας της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ κύριε Χάρπερ. Κύριε Μπούσοϊ, αντιπροσωπεύετε τον κύριο Μάντο σήμερα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ εδώ. Ε, θα ήθελα να παρουσιάσω την άποψή μας για το σημαντικό αυτό φάκελο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Παντσέρη είχε δύσκολο έργο, διότι το θέμα είναι εξαιρετικά τεχνικό και νομίζουμε ότι εκείνος και οι συνάδελφοι σκιώδεις εισηγητές θα μπορέσουν να παρουσιάσουν μια πλήρη έκθεση εφόσον φαίνεται ότι υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων. Πάρα πολλές τροπολογίες που κατατέθηκαν είναι πολύ τεχνικές, αλλά εφόσον εκπροσωπούμε τους λαούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να λάβουμε θέση σχετικά με αυτά τα τεχνικά θέματα. Είμαστε ικανοποιημένοι για το θέμα των οχημάτων παντός εδάφους. Έχουμε ομαδοποίησει τις δυνάμεις μας, τις προσπάθειές μας για μια κοινή θέση. Νομίζω ότι ο εισηγητής και οι σκιώδες θα μπορούν να αναλύσουν ικανοποιητικά για όλους το θέμα αυτών των οχημάτων, όχι μόνο σε αυτή την εισήγηση, αλλά και στην εισήγηση για τα οχήματα της κατηγορίας L πρέπει να διευκρινιστούν ορισμένα θέματα. Ο Τον Μέντερς, ε, ε, η συνεισηγητής, είναι ε, επίσης πεπισμένος ότι χρησιμοποιούνται αγροτικά οχήματα για οδική κατασκευή και θα ήθελε να υπάρχει και μια λύση για το θέμα αυτό επικάλυψη με την οδηγία περί μηχανημάτων θα πρέπει να αποφευχθεί. Ελπίζουμε όλα τα μέρη να μπορέσουν ε, να διαλύσουν τις διαφορές εκεί όπου υπάρχουν. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω το θέμα της χρήσης δημοσίων οδών πρέπει να διευκρινίσουμε τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα αγροτικά και δασικά οχήματα προτού να χρησιμοποιούν τις δημόσιες οδούς. Υπάρχει κάποια διαφορά στα κράτη-μέλη σχετικά με τα διπλώματα οδηγήσεως στις κατοχώρες, Στη χώρα του συναδέλφου των Μέντερς από τα 16 μπορεί κανείς να οδηγήσει ένα αγροτικό ε, όχημα που είναι 10 φορές πιο βαρύ από ένα κανονικό αυτοκίνητο. Θέλουμε να διευκρινιστεί αυτό. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Παντσέρη και την ομάδα του και περιμένουμε ότι θα υπάρξει μια στενή συνεργασία και ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε συνάδελφε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Παντσέρη για την εξαιρετική του δουλειά. Έχω και εγώ... Και εγώ θεωρώ τη δουλειά του εξαιρετική με τις τροπολογίες, ωστόσο υπάρχουν κάποια σημεία ε, τα οποία ανεξάρτητα από αυτά που είπε θα ήθελα να συζητηθούν. Για την κατηγορία L για παράδειγμα, είμαι και εγώ σκιωδής εισηγήτρια για την κατηγορία αυτή και ε, πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Μπούζο σχετικά με τους ε, με το δίπλωμα οδήγηση δεν είναι το θέμα μας πιστεύω αυτή της έκθεσης. Αλλά όταν μιλάμε για τη χρήση σε δρόμου στον ATV, χρειάζεται να βρούμε μία ε, λύση για, την, ε, για το αν θα είναι ή όχι στην κατηγορία L και να δούμε τι γίνεται και με τις εκπομπές καυσαερίων. Και το πρόβλημα λοιπόν που εσείς αναφέρατε, ότι δηλαδή κάποιο ε, στα 16 μπορεί να πάρει δίπλωμα για να οδηγήσει τέτοια μηχανήματα, ε, φυσικά αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε. Φυσικά είναι κάτι το οποίο ε, μας αφορά και, θα, ε, και υπόκειται στην κατηγορία για τους ελκυστήρες και τα δασικά μηχανήματα. Εάν επεξεργαστούμε και, τα, και τους δύο τομείς ταυτόχρονα, τότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και εδώ έχετε δίκιο. Φυσικά πρέπει να προσέξουμε πώς ε, θα το κάνουμε αυτό ταυτόχρονα. Όμως ε, θα ήθελα να παρακαλέσω λοιπόν τον ε, κύριο Παντσέρη να μας βοηθήσει σε αυτό. Κατά τα άλλα υποστηρίζω την δουλειά του κυρίως όσον αφορά την πρόσβαση στις ε, πληροφορίες και, στην, ε, στα εργαστήρια επισκευής των ε, μηχανημάτων αυτών. Και πιστεύω, όπως και ο κύριος Φάμπο, ότι αυτό πρέπει να παραμείνει στην έκθεση. Είναι μια λογική ακολουθία μετά από τις, από τις άλλες ρυθμίσεις. Σας ευχαριστώ κυρία Γούλε. Θα ήθελα να σας ζητήσω... Ε, κύριε Τρεταφυλλίδη, βρίσκεστε, εδώ για αυτό το λόγο. Όχι, είμαι για το επόμενο θέμα. Äh, äh, κύριε Ρώση, βρίσκεστε εδώ στη θέση του κυρίου Σαβίνη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, ναι. Είμαι σκιώδης εισηγητής για τη δική μου ομάδα. Και εγώ ευχαριστώ τον συνάδελφο Παντζέρη για όσα έκανε και για την παρουσίαση που μα έκανε προηγουμένω, καθώ και για την προθυμία του να εξετάσει όλε τι υποβληθεί τροπολογίε. Η πρόταση τη Επιτροπή νομίζω ότι μπορεί να γίνει αποδεκτή, γιατί μπορεί να επικαιροποιήσει και από τεχνική άποψη ε, τι απαιτήσει και επίση ανοίγει την αγορά και σε παραγωγού οχηματών ε, για την συντηρήση. Όμω θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να αποφύγουμε τα προβλήματα για τις παραγωγικές εταιρείες και τους χρήστες των μέσων, των οχημάτων. Θα πρέπει να παρέμβουμε κατά τρόπο ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του προτινόμενου κανονισμού. Το έχω επισημάνει και στον εισηγητή. Κάποιες τροπολογίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές και θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για τη βελτίωση του τελικού κειμένου. Πρώτα απ' όλα Ξέρουμε ότι τα γεωργικά και δασικά οχήματα μπορούν να κυκλοφορήσουν και σε δρόμους, αλλά συνήθως χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά εδάφη, δηλαδή σε γεωργικά ε, εδάφη. Αυτό λοιπόν το θέμα καλύπτεται επαρκώς από την πρόταση της Επιτροπής, καθώς και το ζήτημα της διπλής νομοθέτησης καλύπτεται επαρκώς ε, μέσω της απόκλησης των ελκυστήρων με την οδηγία 2642 για τα γεωργικά οχήματα. Εδώ θα πρέπει να φροντίσουμε βεβαίως να μην συμπέσει η εφαρμογή των κανόνων με τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των κανόνων, των απαιτήσεων που θα προκύπτουν από άλλο ρυθμιστικό πλαίσιο. Δηλαδή, οι ελκυστήρες μπορούν να απολυθούν για την ώρα, χωρί δυσκολίε, αλλά δεν θα πρέπει να εμποδιστεί η πώλησή του από τη διαδικασία ομολογοποίηση που μπορεί μεταξύ να έχει γίνει υποχρεωτική. Θα πρέπει επίση να προσέξουμε τι θα γίνει με τι εφαρμοστικέ πράξει και τι κατεχώρηση πράξει που θα προβληθούν και την, ε, το κατά πόσο θα είναι υλοποιήσιμε. Δηλαδή, σε ποιο χρόνο θα επιβάλλουμε απαιτήσει στου παραγωγού. Για τι τεχνικέ προδιαγραφέ επίση που θα αναλάβουν οι κατασκευαστέ, όλα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν εφόσον οι ε, γεωργοί ξέρουμε ότι χρησιμοποιούν ε, τα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση αντικτύπου σε κάθε περίπτωση εδώ και να λάβουμε υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των ε, διαφορών οχημάτων. Θα πρέπει ήδη από τον κανονισμό να έχουμε ορίσει διαδικασίες ομοιογενείς για τις διαδικασίες που θα εφαρμόζονται για τους κατασκευαστές επειδή υπάρχουν εκατοντάδε τύποι οχημάτων και μεγάλη ποικιλία στην αγορά, θα πρέπει παραγωγή να ε, γνωρίζουν για ποιους σκοπούς θα κατασκευάζουν και με βάση τι απαιτήσει τα οχήματα, τα οποία μπορεί να είναι εμπορικά ή όχι. Και υπάρχει από τη μια το δικαίωμα των μικρών παραγωγών, αλλά και των πολιτών που θα χρησιμοποιούν τα οχήματα να απευθύνονται σε κέντρα βοήθεια, σε ειδικά κέντρα. Να προσέξουμε να μην δημιουργήσουμε εδώ μεγάλα προβλήματα. Επίση, η συμπερίληψη τη κατηγορία U τον κανονισμό. Εδώ μιλάμε για κινητά, κινητά οχήματα, ιδιαίτερα περίπλοκα, με περιορισμένο αριθμό μάλλον, και από την άποψη της ασφάλειας και από την άποψη του περιβαλλοντικού του αντικτύπου. Εδώ πάντως συμφωνούμε με την πρόταση του συγητή ότι θα πρέπει να εναρμονιστεί το θέμα των μηχανημάτων, των κινητών ε, μηχανημάτων, γιατί ανάλογα με τους κανόνες οδικής ασφάλειας διαφέρουν ε, οι ρυθμίσεις και απαιτήσει από κράτος σε κράτος. Θα πρέπει εδώ λοιπόν η οδική κυκλοφορία να εναρμονιστεί μεταξύ των κρατών μελών. Εύχομαι με την τεχνική συνάντηση που θα έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα, την ε, Δευτέρα και μετά στην επόμενη συνάντηση με τους κόδους εισηγητές, να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που να, πετύχει σχεδόν τη συνένεση όλων των ενδιαφερόμενων. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας έδωσα το λόγο για λίγο παραπάνω. Πρέπει όμως να προσέξουμε το χρονοδιάγραμμά μα. Δεν υπάρχουν άλλες τοποθετήσει για άλλα μέλη. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Ζων, αν θέλετε μπορείτε να πάρετε το λόγο. Και προσέξτε παρακαλώ το χρόνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μελετήσαμε με ιδιαίτερη προσοχή την έκθεση του κυρίου Παντζέρη και θεωρούμε ότι είναι μια έκθεση ποιοτική. Μια συμβολή που θα μας είναι χρήσιμη για την εξακολούθηση των εργασιών μας. Συνειδητοποιούμε ότι το θέμα είναι άκρως τεχνικό. Όμως για όλα τα επί της ουσίας ζητήματα, οι παρατηρήσεις και οι συνεισφορές του κ. Παντζέρη ανταποκρίνονται ακριβώς αυτό που και εμείς επιζητούσαμε. Να απλουστεύσουμε την νομοθεσία δηλαδή και να την καταστήσουμε αποτελεσματική και για τους ε, ενδιαφερομένους τους μετέχοντες της αγοράς. Τρία είναι τα ζητήματα που μας ενδιαφέρουν κυρίως και για εμά. Πρώτον, το πεδίο εφαρμογή του κειμένου, διότι η ισχύουσα κατάσταση δεν ήταν ικανοποιητική. Υπήρχαν διαφορετικέ υποχρεώσει για διαφορετικέ κατηγορίε, μια σειρά από διαφορετικέ κατηγορίε οχημάτων. Προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε το σύνολο των υποχρεώσεων πιο ομοιογενέ. Όμω, εδώ έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία να γίνει ακόμη πιο ομοιογενέ το σύνολο. Το Κοινοβούλιο θα αποφανθεί περίπου ταυτόχρονα για τους ελκυστήρες και την κατηγορία L, και ε, αυτό είναι μια πολύ καλή περίπτωση για να προχωρήσουμε ως προς την συνέπεια και το τι καλύπτει το αρχικό κείμενο. Δηλαδή την ομοιογένεια των υποχρεώσεων. Εδώ, για τις επισκευές και τη συντήρηση, τις σχετικές υποχρεώσεις, καταλαβαίνουμε ότι ο εισηγητής αναζητά την ισορροπία μεταξύ αυτών των υποχρεώσεων που επιτρέπουν στους ανεξάρτητους ε, επισκευαστές να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και μετά ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα καθώς και ταυτόχρονα την υποχρέωση σεβασμού των ε, δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία που διαφέρουν από όχημα σε όχημα και από κατηγορία σε κατηγορία. Ιδιαίτερα προσφυλή μα είναι τα σχόλια του εισηγητή για τον τρόπο που θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τα δεδομένα, την ε, αποστολή δεδομένων για του επισκευαστέ. Μετά, το τρίτο θέμα είναι η ημερομηνία θέση σε ισχύ. Ξέρετε ότι δεν είμαστε σχολαστικοί ω προ το θέμα αυτό. Θα πρέπει να βρούμε μια λύση ρεαλιστική που να λαμβάνει υπόψη και την ταχύτητα με την οποία θα προετοιμαστούν ε, οι εφαρμοστικέ πράξει ή η κατεχώρηση πράξη. Δηλαδή, για ένα έργο τόσο περίπλοκο και για τόσα πράγματα που μένουν να γίνουν, θα πρέπει να βρούμε μια τέτοια λύση ώστε να είναι η ημερομηνία θέση σε ισχύ πραγματιστική. Να μπορέσουν ε, ε, εγκαίρω να προετοιμαστούν και οι κατακρουσιοδότηση πράξεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν πραγματικά περιεκτικός, σύντομος και ξεκάθαρος. Αγαπητέ κύριε Παντσέρη, θα θέλατε να πείτε κάποια τελευταία λόγια. Παρακαλώ, σας ακούω. Grazie. Ευχαριστούμε. Ένα λεπτό θα χρειαστώ. Να πω ότι νομίζω τρία είναι τα ζητήματα στα οποία πρέπει να επικεντρωθούμε την ερχόμενη εβδομάδα, από ό,τι καταλαβαίνω. Και ελπίζω και από τη συζήτησή μας να προκύψουν οι κατάλληλες συμβαστικέ λύσεις. Πρώτον, η πρόσβαση στις πληροφορίες. Εδώ νομίζω ότι μπορούμε ήρεμα να το μελετήσουμε, ώστε να ανταποκρίνονται μεταξύ τους οι διάφορες υποχρεώσεις και απαιτήσει. Δεύτερον, η θέση σε ισχύ. Η προσέγγιση μου ταυτίζεται με αυτήν τη Επιτροπή. Θέλουμε να είμαστε ρεαλιστέ, λαμβάνοντα υπόψη τι απαιτήσει των παραγωγών και το γεγονό ότι μπορεί να υπάρχει επικάλυψη νομοθετικών υποχρεώσεων. Αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να εξεύρουμε λύσει. Το ίδιο σκόπιμο θα ήταν να γίνει μια περαιτέρω συζήτηση για το θέμα των κατηγοριών, της κατηγορίας των ATV μάλλον, των επαγγελματικών οχημάτων παντός εδάφους, ώστε η συνολική λύση να συγκεντρώνει την ευρύτερη δυνατή συνένεση. Εγώ είμαι διαθέσιμος να γίνουν όλες οι σχετικές συζητήσεις και ελπίζω να καταφέρουμε να συγκλίνουν όσο το δυνατόν περισσότερες ε, απόψεις από του συναδέλφου βουλευτέ και του κοιόδη εξηγητέ. Για ένα θέμα που, όπω σωστά είπατε, είναι τόσο σημαντικό όχι μόνο από τεχνική άποψη, αλλά και των εκθέσεων του Κοινοβουλίου που καθορίζουν το μέλλον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνιο, για την δουλειά που κάνει, που μπορεί να ακούγεται πολυτεχνική. Έχει όμως εξαιρετικά μεγάλη πολιτική σημασία. Η έκθεση είναι πολύτιμη. Να σας υπενθυμίσω, η ψηφοφορία είναι στις 5 Δεκεμβρίου, για τότε προβλέπετε, στην Επιτροπή και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια, Ολομέλεια μάλλον το Φεβρουάριο του 2012. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παντσέρη. Λοιπόν, τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Η έκθεση του Λουιγκρέχ για την ε, Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια 2010, αποδομώντα τα εμπόδια για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα θα λάβω ρόλο συντονίστριας, θα περνώ από, τον, από τη μία αρμοδιότητα στην άλλη. Δυστυχώ ο κύριος Γκρέκ είναι άρρωστο και δεν μπορεί να έρθει εδώ και μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω, γιατί είναι σημαντικό να προχωρήσουμε με τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να σας το παρουσιάσω σύντομα. Ο κύριος Γκρέκ έχει κάνει κάποιες ε, παρατηρήσεις. Θα ήθελε να ε, τονίσει ότι φυσικά αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες να φέρει σε αυτό το κείμενο να, να, όλα όσα χρειάζονται, όλα όσα ήταν αναγκαία να υπάρχουν σε αυτό το κείμενο. Προσπάθησε να μην ξεπεράσει τα όρια που είχε και φυσικά συνάντησε ε, πολλά προβλήματα γιατί αυτά τα θέματα είναι εκτενέστατα, πολύ σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την κοινωνία των πολιτών της. Ε, και, αλλά προσπάθησε να επικεντρωθεί στις αρμοδιότητες της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ και αυτές να παρουσιάσει σε αυτή την έκθεση. Και πράγματι, ο ορισμός της ε, ηθαγένειας του Ευρωπαίου πολίτη καλύπτει πολλούς ε, τομείς. Ε, έχει να κάνει με πολλές εθνικές ταυτότητες, έχει να κάνει με φοιτητέ, με επαγγελματίε, με καταναλωτές, με απλούς πολίτες, με εργοδότες, με εργαζόμενους κτλ. κτλ, κτλ. Πολλοί είναι οι ρόλοι, πολλούς καλύπτει αυτή η έκθεση. Και όταν μιλάμε για πολίτες της Ευρώπης έχουμε να κάνουμε με όλα αυτά. Αυτό λοιπόν ήταν ένα πολύ σημαντικό έργο και πρέπει να δούμε περί τίνος πρόκειται. Ο κύριος Γκρέχ επίσης θεωρεί, θεωρεί πολύ σημαντικό το ερώτημα ποιος, τι είναι η ευρωπαϊκή ηθαγένεια ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων γνωρίζει λίγο πολύ ότι η ευρωπαϊκή ηθαγένεια είναι κάτι που υπάρχει, είναι κάτι το απτό και μόνο το 1 τρίτο των ε, ανθρώπων όμως γνωρίζουν ή τουλάχιστον θεωρούν πως γνωρίζουν ότι έχουν δικαιώματα ως Ευρωπαίοι πολίτες, ως πολίτες της Ένωσης. Και αυτά τα νούμερα είναι εκπληκτικά. Διότι από το 1994 θα έπρεπε να είναι ίσως λίγο περισσότερα τα, το ποσοστό των ανθρώπων που είναι ενημερωμένοι. Οι τομείς, όπως προείπα, είναι Πολύ και διαφορετική Είναι η οικονομική ολοκλήρωση των πολιτών, η κοινωνική ολοκλήρωση σε μία σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και όσο το δυνατόν χωρίς ε, σύνορα. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο κύριος Γκρέκ προσπάθησε να ε, συνδέσει τις διαφορετικές συμβουλευτικές έρευνες και μελέτες από τα διαφορετικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τη συνδέσει στην δική του έκθεση. Θεωρεί πως είναι καιρός για τους πολίτες να έρθουν στο προσκήνιο της ε, πολιτικής πραγματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουν πλήρη, αντίληψη των, ε, της ευρωπαϊκής τους ιδιότητας. Μα συγχωρείτε γιατί έχει γράψει τα αγγλικά και η μετάφραση, η μετάφρασή μου είναι λίγο πρόχειρη και λίγο ελεύθερη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, εκτός από τον παραδοσιακό ορισμό του Ευρωπαίου πολίτη, να αναλογιστούμε ε, αυτήν την νέα προσέγγιση σε αυτό το επίπεδο. Η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη είναι κάτι που πρέπει να ε, σκεφτούμε, πρέπει να εμβαθύνουμε και αυτό είναι κάτι που έχει ήδη γίνει μία φορά. Και ε, είναι κάτι το οποίο έχει ε, λάβει και δημοσιότητα, είναι κάτι το οποίο ο κύριος Μάριο Μόντι συμπεριέλαβε στο έργο του. Προς το παρόν, η μελέτη της Κομισιόν για, την, για το Consumer Empowerment έχει δείξει ότι η εφαρμογή του δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαφέρει πάρα πολύ από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν διαφορετικές ε, νομοθετικές εργασίες και αυτό σημαίνει διαφορετικά προβλήματα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα για εκείνους που ε, διαμένουν σε παραπάνω από μία ε, χώρα ή που μετακινούνται μεταξύ των ε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο τα σύνορα που, της εσωτερικής αγοράς να καταργηθούν και να καταργούνται σταδιακά έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ελεύθερη μετακίνηση των ε, προσώπων, των αγαθών, των υπηρεσιών και του κεφαλαίου. Και με τον τρόπο αυτό οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να, να καταφέρουν να κερδίσουν ε, εμπιστοσύνη στις αγορές. Και αυτό θα γίνει εφόσον οι πολίτες είναι σωστά και πλήρως ενημερωμένοι. Αυτό θα τους φέρει πολλά πλέον και θα τους δώσει πολλά δικαιώματα τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν. Γι' αυτό λοιπόν η πληροφορία είναι πολύ βασικό σημείο. Το πιο σημαντικό σημείο πρέπει να είναι στο κέντρο των προσπαθειών μας. Και, δεν, και πρέπει να προσέξουμε να μην δώσουμε στους πολίτες έναν πακτολό πληροφοριών που δεν είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους και έτσι ώστε και εκείνοι να μην μπορούν να διαλέξουν, να, να ξεχωρίσουν. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες για τους ε, πολίτες. Τόσες πολλές όμως, τόσο πολύπλοκες και τόσο ασυντόνιστες ώστε οι πολίτες οδηγούνται σε σύγχυση και δεν θα μπορούν να διακρίνουν το σημαντικό από το λιγότερο σημαντικό. Όσον αφορά τους ε, καταναλωτές και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τώρα, θα πρέπει να ε, προσέξουμε να βρεθούν μηχανισμοί ADR ε, εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών και επίσης να γνωρίζουμε ότι και η Κομισιόν θα έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί με αυτό και να βελτιώσει τους ε, μηχανισμούς αυτούς ADR. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό όχι μόνο να έχουμε ένα σωστό ε, σύστημα ADR, αλλά και να το έχουμε από το 2012. Να το φροντίσει αυτό η Κομισιό. Ο κύριος Γκρέκ τέλος ελπίζει ότι θα υπάρξει μια καλή συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές ότι οι τοποθετήσεις θα είναι παραγωγικές και ελπίζει τέλος σε μια πολύ ε, θετική συνεργασία ανάμεσα στους ε, σκιώδεις εισηγητέ. Και τώρα επανέρχομαι στο ρόλο μου ως πρόεδρος ε, αυτής της Επιτροπής και θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σάιμον Μπουσουτήλ ως εκπρόσωπο, ως σκιώδη εισηγητή του ΕΛΚ. Σάιμον, έχετε το λόγο. Eh, eh, eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου προς τον κύριο Γκρέκ. Νομίζω ε, είναι άρρωστος, γι' αυτό δεν μπόρεσε να είναι εδώ μεταξύ μας. Ελπίζω να αναρρώσει σύντομα. Θα ήθελα να τον συγχαρώ για αυτή την εισήγηση που είναι για ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει όλους και θα πρέπει ε, να έχει μεγάλη υποστήριξη διότι ο στόχος της έκθεσης αυτής είναι κάτι για το οποίο όλοι συμφωνούμε. Η σημασία να άρουμε όλα τα εμπόδια στα οποία προσκρούν οι πολίτες όταν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις κανονισμούς της εσωτερικής αγοράς και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Ο κύριος Γκρέγκα επισημαίνει ε, δύο βασικά θέματα. Πρώτα απ' όλα Έχουμε την, ε, ε, την, τα ψηφίσματα εναλλακτικών ε, διαφορών, ρύθμιση διαφορών και νομίζω ότι αυτό το σύστημα, το ADI, είναι ένα πολύ καλό σύστημα, είναι χαμηλού κόστους και μπορεί κανείς να διευθετήσει τις διαφορές και ο κύριος Γκρέχα επισημαίνει με λεπτομέρειες την σημασία τα δικαιώματα πληροφόρησης, ενημέρωσης των πολιτών. Πρέπει να μπορούν να ασκήσουν αυτά τα δικαιώματα. Επίσης, χαίρομαι που συνεργάζομαι με τον κύριο Γκρέκ για το θέμα αυτό, όχι μόνο επειδή θα ε, ήταν ικανοποιημένος που μπορώ να μιλήσω στην μητρική μου γλώσσα, αλλά επειδή και συμβάλλω σε μια εισήγηση την οποία εκείνος συμπλήρωσε. Ε, ε, για μια άλλη έκθεση. Έχουν αρχίσει συζητήσεις ε, αυτήν την εβδομάδα, τη Δευτέρα. Ήσασταν παρούσα, κυρία Πρόεδρε, όταν είχαμε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την έκθεση που θα οργανώσω εγώ για τον πίνακα βαθμολόγησης εσωτερικής αγοράς, για το scoreboard. Αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στο θέμα αυτό. Σχετικά με τι τροπολογίε. θα παρουσιάσω έναν ορισμένο αριθμό τροπολογιών ούτως ώστε να τονίσω περισσότερο την ανάγκη να τονιστεί ακόμα περισσότερο το θέμα των λύσεων. Είναι κρίσιμο να ξέρουμε ότι όταν ξέρουμε τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι πολίτες να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην εξέβρεση λύσεων, των λύσεων που απαιτούνται. Επιπλέον θα ήθελα να τονίσω ότι η Επίτροπη όχι μόνο εργάζεται για νέα νομοθετήματα και μελέτες, αλλά θέλει να βεβαιωθεί ότι είναι πιο αποτελεσματική και αποφασιστική στην εφαρμογή των αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί. Νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι ότι αυτό που ήδη υπάρχει να μπορεί να, μπορεί να αποδώσει τους περισσότερους δυνατούς καρπούς και ωφέλη. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω δεν ε, θα ήθελα να μακρηγορήσω στην ε, παρέμβασή μου, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι ελπίζω ο κύριος Γκρέγκ και εγώ θα μπορέσουμε ε, να έχουμε συμβιβασμό, συμβιβασμούς με τις τροπολογίες και να συμφωνήσουμε για αυτή την εισήγηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. και Μπουσό, έχετε το λόγο όχι ω εκπρόσωπος αλλά ω πραγματικά ισχυώδης εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκρέχ για τις προσπάθειες που έκανε να συντάξει το σχέδιο της έκθεση αυτής ε, για το φόρουμ τη ενιαίας αγοράς. Και ακούσαμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτε ε, όσον αφορά την ενιαία αγορά, την εσωτερική αγορά. Φυσικά δεν μπορούσαμε να βάλουμε τα πάντα στο σχέδιο της ε, γνωμοδότησης, όμως πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες ε, καλές ιδέες και αξίζει να τις υποστηρίξουμε. Σίγουρα υπάρχουν κάποια φράγματα στην ελεύθερη μετακίνηση των προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου και πραγματικά ε, αυτά τα προβλήματα αποτελούν εμπόδιο στην ενιαία αγορά και παρεμποδίζουν την κινητικότητα. Ο κύριος Γκρέκ έχει δίκιο ότι οι πολίτες, ε, λέγοντας ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους και ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ε, ε, οφείλονται σε έλλειψη παρκών πληροφοριών. Φυσικά χρειάζεται να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Υπάρχουν όμως κάποια δικαιώματα τα οποία οι πολίτες τα έχουν υπόψη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πληροφορήσουμε και να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες και να τους πληροφορήσουμε για τα δικαιώματά τους και για τις, ε, για τις υποχρεώσεις τους και για τις συνθήκες ε, στις οποίες ζουν. Αρκετοί πολίτες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην, ε, στο μητρό ε, αυτοκινήτων όταν αγοράζουν αυτοκίνητο από κάποιο άλλο κράτος μέλος. Και πιστεύουμε λοιπόν ότι η άρση των φραγμάτων θα επιλύσει το πρόβλημα αυτό. Επίση, υπάρχουν πολίτε που έχουν πρόβλημα να ανοίξουν τραπεζικού λογαριασμού σε κάποιο άλλο κράτο μέλο αρκετοί πολίτες ε, αποκλείονται οικονομικά και δεν έχουν βασικούς ε, ε, τραπεζικούς λογαριασμούς πληρωμών. Έτσι λοιπόν για να αυξήσουμε την κινητικότητα πρέπει σίγουρα να διευκολύνουμε την πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα από το ένα κράτος στο άλλο. Επίσης πρέπει να δώσω έμφαση στην διαφάνεια, στην έννοια της διαφάνειας για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο τραπεζικό σύστημα. Επιπλέον, μόνο Επιπλέον, έχουμε υιοθετήσει μια οδηγία για την καλύτερη πληροφόρηση των ε, πολιτών και ιδιαίτερα για το κόστος των ε, τραπεζικών λογαριασμών. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ε, του ενημερώσουμε περισσότερο, επίση και στον τομέα τη υγειονομική περίθαλψης και πάνω στα δικαιώματά του γι' αυτό. Έπειτα, μιλήσαμε για του μηχανισμού ADR, επίλυση ε, διαφορών. Αυτά είναι σημαντικά εργαλεία για του πολίτε. Ε, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα δικαιώματά του και οι μηχανισμοί αυτοί είναι πιο, ε, πιο φτηνοί. Όμω πρέπει να του ενημερώσουμε για το πώ μπορούν να του χρησιμοποιήσουν. Και αυτή είναι μια σημαντική άποψη και, μια, και ένα σημαντικό τομέα στον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Έχετε θέσει ορισμένα σημαντικά σημεία. Ε, βλέπω ότι δεν είναι εδώ ούτε η πράσινη ούτε η συντηρητική. Κυριάκο, λοιπόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ τον Λούι Γκρέχ για την εργασία που έχει παρουσιάσει και να συμφωνήσω μαζί του πάνω σε πολλά από τα σημεία τα οποία αναφέρει, όπως για παράδειγμα ότι υπάρχει ανάγκη να παραμεριστούν τα εμπόδια τα οποία έχουν ε, εντοπιστεί και που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε διάφορους ε, τομείς, όπως είναι το εμπόδιο της ελεύθερης κυκλοφορίας, για παράδειγμα. Ε, τα εμπόδια που, στα οποία γίνονται αναφορές σε ορισμένα κράτη-μέλη, όπως είναι η αναγνώριση πλήρως των δικαιωμάτων των μελών οικογενειών που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών για έκδοση αδειών παραμονής περιορισμένης διάρκειας. Άλλα θέματα είναι επίσης οι δυσκολίες όσον αφορά την ανανέωση των ταξιδιωτικών τους εγγράφων, δυσκολίες σε σχέση με την πρόσβαση στα δικαιώματα τους στην κοινωνική ασφάλιση, όπως επίσης όσον αφορά την άρνηση κυβερνήσεων να χορηγήσουν παροχές όπως το επίδομα διαβίωσης αναπήρου, το επίδομα βοηθείας, το επίδομα επιμελητή αναπήρου. Επίσης προβλήματα που αφορούν την αναγνώριση τίτλων σπουδών ή προσόντων και η ανεπαρκή μεταφορά ή εφαρμογή της Οδηγίας 2005-36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέλος, ζητήματα φορολογίας θέτουν σημαντικά εμπόδια στην άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας. Για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο μπορεί να φορολογείται σε διάφορες χώρες εάν υπάρξουν διαδοχικές αλλαγές του τόπου κατοικίας. Όλα αυτά παρουσιάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως κατακαιρματισμένη. Ο κατακαιρματισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως αποδίδεται στην έλλειψη ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι υπάρχουν και άλλοι, λόγοι εξίσου ισχυροί όπως η ύπαρξη μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικών ταχυτήτων στην ανάπτυξη, την οικονομική ευρωστία κλπ. Η γνωμοδότηση επίσης προβάλλει την άποψη ότι το πρόβλημα της οικονομικής ολοκλήρωσης που θα έχει ως συνέπεια την ενίσχυση της θέσης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δημιουργία μιας νέας πολιτικής όθησης στην έννοια της ιδιότητας του πολίτη θα επιτευχθεί μέσω της ενιαίας αγοράς. Εμείς προσθέτουμε πως ναι, αυτό μπορεί να γίνει μέσω μιας ενιαίας αγοράς που θα σέβεται τους εργαζόμενους και το περιβάλλον και ότι η πραγματικά σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων είναι που θα φέρει τη βιωσιμότητα και που ενισχύει την ιδιότητα του πολίτη. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα υποβάλουμε τροπολογίες και θα συνεργαστούμε με τον Λούιν Κρέχ για να περάσουμε αυτά τα μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις από τους συναδέλφους, ε, αν όχι και φαίνεται πως όχι, τότε κυρία Κιαραντάμο, θα θέλετε να μας, να μας πείτε δύο λόγια. Έχετε το λόγο. Thank you, Ευχαριστώ. κυρία Πρόεδρε. Από πλευράς της Επιτροπής θέλω να χαιρετήσω το σχέδιο έκθεσης τη συμβολή για αυτήν την έκθεση και τονίζει την συμπληρωματικότητα ε, με ε, συμπληρωματικές εργασίες ε, όπως την πράξη για την ενία αγορά. Θέλουμε την άρση των εμποδίων που συναντούν οι πολίτες όταν ασκούν τα στην καθημερινή ζωή, όταν ε, ασκούν τα δικαιώματά τους βάσει της συνθήκης και τα δικαιώματα ελεύθερης διακίνησης. Είναι σημαντικό να έχουμε μια τέτοια συζήτηση, έκθεση προσδιορίζει 25 δράσεις για να αρθούν τα εμπόδια αυτά. Πολλές από τις δράσεις αυτές αναφέρθηκαν από τα μέλη, όπως τα αυτοκίνητα, όπως η εναλλακτική ε, διευθέτηση διαφθορών και νομίζω ότι η έκθεση Γκρέκ είναι αξιοσημείωτη σχετικά με τις δράσεις. Νομίζω ότι η εναλλακτική διευθέτηση διαφορών έχει εξέχουσα θέση στην έκθεση και νομίζω ότι και η Κομισιόν θα κάνει ε, μια πρόταση για μια οδηγία σχετικά με αυτήν την διευθέτηση διαφορών και μια άλλη οδηγία. Επίσης εργαζόμαστε για την ε, επιβολή για την υλοποίηση μιας οδηγίας. Η υλοποίηση αναφέρθηκε από διάφορους βουλευτές, ευρωβουλευτές και ε, νομίζω ότι στα συμπεράσματα η Επιτροπή συμπεραίνει ότι μεταξύ των εμποδίων αυτών και των δράσεων των μέτρων για να επιληθούν η σημαντικότερη δράση που πρέπει να αναλυφθεί δεν είναι οπωσδήποτε νέα νομοθεσία αλλά σωστή εφαρμογή από τα κράτη-μέλη των υφισταμένων κανόνων και η Επιτροπή εφαρμόζει ε, τα, τα νομοθετήματα και αποδίδει προτεραιότητα σε πάρα πολλούς τομείς όπως είναι η ελεύθερη διακίνηση ατόμων και οι διαδικασίες επί παραβάση κατά τη διάρκεια των έξι τελευταίων μηνών. Παρακολουθούμε επίσης τα ε, συμπεράσματα του Κράκολ που νομίζω ότι συμπίπτουν με τις προγενέστερα συμπεράσματα. Η ε, σημασία του Σολβίτ και των ε, κέντρων που βοηθούν τους ε, πολίτες και η ανάγκη για μια πιο συντονισμένη δράση νομίζω ότι είναι σημαντικό. Η Κομισιόν επίσης μιλάει για την ανάγκη να υπάρχει μία μόνο θηρίδα εξυπηρέτησης και να μην υπάρχουν 15 ας πούμε, ε, η δίκτυα καταναλωτών, το, η Solvita, ε, θα πρέπει ε, να, να, να κατευθύνονται οι πολίτες προς το πιο, την πιο κατάλληλη θηρίδα, το πιο, το πιο κατάλληλη υπηρεσία για να επιλύσει το πρόβλημά του. Θα έχουμε ένα εγχειρίδιο στο τέλος του έτους που σε όλες τις γλώσσες ε, αυτό, αν θέλετε, το εγχειρίδιο, το εικονικό για ε, τους ε, πολίτες που αναφέρεται στην έκθεση Greg. Επίσης, η ευαισθητοποίηση αναφέρεται και μία από τα μέτρα σε αυτήν την έκθεση είναι να έχουμε την Ευρωπαϊκό Έτος του Πολίτη. Αυτή έθηκε και συζητείται Παράλληλα και εδώ και στο Συμβούλιο η Επιτροπή πιστεύει ότι θα υπάρξει υποστήριξη για αυτή την πρόταση, ούτω ώστε να αυξήσουμε αυτήν την συνειδητοποίηση. Νομίζω ότι η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών έχουν ε, μάθει για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια, ε, πάνω από 80%, αλλά μόνο 43% ξέρουν περί τίνος πρόκειται σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση την οποία είχαμε. Ε, θα, σίγουρα θα μεταβιβάσουμε στον κύριο Γκρέκ τα όσα υπόθηκαν σήμερα. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι του χρόνου έχουμε τα 20 χρόνια νέας αγοράς. Είναι κάτι που θα γιορτάσουμε και ε, πρέπει να το λάβουμε υπόψη και να ε, συνειδητοποιούμε ότι αυτή η εσωτερική αγορά είναι για τους πολίτες. Και ε, αυτό πρέπει να συνδέσει και την ε, αναφορά. Κύριε Μπουσουτήλ, σας ακούσαμε. Υπάρχει επίση η έκθεση για του τραπεζικού λογαριασμού και υπάρχουν όλα αυτά τα, τα πράγματα τα οποία είναι εξαιρετική σημασία για του πολίτε. Και σκέφτομαι ε, ε, ότι εάν καταφέρουμε να το επιτύχουμε αυτό ε, την επόμενη χρονιά, θα μπορέσουμε να δείξουμε στου πολίτε ότι η ενιαία αγορά είναι για εκείνου και εάν το καταφέρουμε αυτό, θα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα την χαίνει μεγαλύτερη αποδοχή από του πολίτε. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που παρευρεθήκατε εδώ Η προθεσμία για τροπολογίε είναι 29 Νοεμβρίου στι 12 το μεσημέρι. Όπως πάντα, το γνωρίζετε, στις 20 Δεκεμβρίου θα εξετάσουμε και θα συζητήσουμε τις ε, τροπολογίε στην Επιτροπή και η ψηφοφορία προβλέπεται επίσης για τις 20 Δεκεμβρίου. Η κύρια Επιτροπή θα ψηφίσει στις 13 Ιανουαρίου, γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να έχουμε τελειώσει τις εργασίες μας πριν από αυτό. Και η, η ψηφοφορία της έκθεσης αυτής προβλέπεται για την Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Είμαι σίγουρη ότι ο κύριος Γκρέιχ θα συνεχίσει να εργάζεται για αυτή την έκθεση και είμαι σίγουρη πως ε, θα σας, ε, σας ευχαριστεί όλους για τη συνεργασία σας, όλους τους σκιώδεις εισηγητές και τώρα θα προχωρήσω στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, τα διάφορα. Δεν έχω κάτι να πω, εάν εσείς έχετε κάτι να πείτε τότε... Ε, πείτε το αλλιώς έχουμε τελειώσει. Το μόνο που μένει να πω είναι ότι η επόμενη συνεδρίασή μας θα λάβει χώρα την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου και μετά από αυτό σας εύχομαι καλή επιστροφή στα σπίτια σας ε, και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.